Dear colleagues, could you please take seat? We open... Ο Πρόεδρος, καθίστε παρακαλώ. Άρχεται η συνεδρίαση. Και καλώς ορίσατε. Έχουμε το σημείο υπαριθμών 10 της ημερησίας διατάξεως. Καλώς ορίσατε τον Τζον Μπέργαν, ο οποίος είναι ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ε, Αρμόδιας Γενικής Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΟΠΑ ε, ο διοικητής ο κύριος ε, Μπερναρντίνο για δεύτερη μέρα και όπως τα γνωρίζουν οι αγαπητοί συνάδελφοι τώρα θα συζητήσουμε ένα σημαντικό θέμα που είναι ο κατεξουδότηση κανονισμός που αφορά τα έγγραφα με σημαντικές πληροφορίες, το PRIPS. Έχετε λάβει τα σχετικά έγγραφα. Ο διάλογος ήταν εντατικός όσον αφορά την θέση ισχύ του PRIPS θεωρεί το Κοινοβούλιο ότι το ΠΡΙΠΣ και τα σχετικά πληροφορικά έγγραφα είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για περισσότερη διαφάνεια και προστασία των καταναλωτών. Περιτεύει να σα υπενθυμίσω ότι έχουμε ανταλλάξει επιστολέ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεκινήσαμε Φεβρουάριο και Μάρτιο τότε. Επεσήμενε το Κοινοβούλιο κάποια προβλήματα. Μας ε, Απήντησε ο Λορδός Χιλ, κατόπιν συνεχίστηκε ο διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν απευθύναμε άλλη επιστολή πριν τη θέση σε ισχύ του κανονισμού και εκεί επισημάνομαι τι μας προβληματίζει. Δυστυχώς, ο κανονισμός, όπως τα βλέπει η Επιτροπή μας, δεν μας ικανοποιεί, δεν καλύπτει τις ανησυχίες μας και γι' αυτό το καλοκαίρι πολλές πολιτικές ομάδες υπέβαλαν τις ενστάσεις Ανέλαβε ο εισηγητής ο οποίος θα λάβει το λόγο και θα μας τα εξηγήσει καλύτερα. Αυτό είναι μια σημαντική αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το να υποβάλει ένσταση για κάποια κατεξοδότηση πράξη. Οπότε επικαλείται αυτή την αρμοδιότητα το Κοινοβούλιο. Οι λόγοι είναι και διαδικαστικοί. Ότι δηλαδή οι αρχικές αντιρρήσεις του Κοινοβουλίου δεν καλύφθηκαν. Αλλά δεν είναι μόνο διαδικαστικοί οι λόγοι, είναι και λόγοι ουσίας. Έχουμε δύο βασικά προβλήματα με το κείμενο το οποίο σήμερα θα ψηφίσουμε. Πρώτα-πρώτα τις δίκαιες συνθήκες ε, ανταγωνισμού, μεταξύ δηλαδή των ε, διαφορετικών προϊόντων που προσφέρονται. Και το άλλο πρόβλημα είναι ο υπολογισμός των αποδόσεων και επιδόσεων. Θα σας τα πει όμως καλύτερα ο συγητής. πολύ σημαντικό θέμα αυτό, θα τα πούμε πριν την ψηφορία. και δούμε τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΟΠΑ. Τώρα η συγγήτρια θα λάβει το λόγο υπερβόνς Μπερές και κατόπιν να μας πούνε τη γνώμη τους τα πολιτικές ομάδες, κατόπιν η κύριε Μπερναρντίνο και ο άλλος κύριος Μπερναρντίνος. Πρόεδρε, ευχαριστώ, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΙΟΠΑ προς την ανταλλαγή απόψεων. Αρχίσαμε επομένως την συζήτηση για τις ε, αντιρρήσεις μας. Πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία. Θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Και δεν χρειάζεται να ξαναπούμε πόσο σημαντικό νομοθέτημα είναι το PRIPS. Σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό θα πρέπει οι προσφέροντες κάποια συγκεκριμένα προϊόντα να έχουν διαθέσιμα κάποια σημαντικά ενημερωτικά σημειώματα ή έγγραφα για τους ε, επενδυτές λιανικού επίπεδου. Δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα αυτό το έγγραφο απλώς. Αυτός ο μικροεπενδυτής θα πρέπει να είναι να συγκρίνει τα διάφορα προϊόντα για να μπορεί να κάνει την καλύτερη επενδυτική κίνηση. Θα πρέπει λοιπόν να εντάσσεται στη λογική της ιστορικής ενίας αγοράς και να προστατεύει τον καταναλωτή. Στο πρώτο επίπεδο είχαμε ευρύτατη πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο. 637 βουλευτές, μόλις 26 ήταν κατά και 16 αποχές σε σχέση με το κείμενο. Μα συνένωσε επομένω αυτή η ψηφοφορία και αυτό δείχνει πόσο σημαντική θεωρούμε την ελόγω νομοθεσία. Έχουμε επομένω τρεις ε, αντιρρήσεις που προέκυψαν από ε, αυτά που μας αποσχολούν δηλαδή για το RTS, για αυτά τα μέτρα που θέλουμε. Πρώτα-πρώτα υπάρχει μια ένσταση θεσμική. Εμείς προσπαθήσαμε για να έχουμε ε, κατοχυρωμένα κάποια δικαιώματα στο δεύτερο επίπεδο. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντική η πανέβαση του Κοινοβουλίου από πλευράς δημοκρατικής λειτουργίας, από πλευράς εφαρμογής της νομοθεσίας όταν έρθει η ώρα. Εδώ παίξαμε λίγο κρυφτούλιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν είναι ότι δεν θέλουμε καθόλου το ΕΡΤΕΣ. Απλώς θέσαμε κάποια ερωτήματα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέχισε στη δημοσιοποίηση, δημοσίευση του ΕΡΤΕΣ χωρίς να μας καλύψει. Πρόκειται για αυτά τα μέτρα δευτέρου επίπεδου. Έχω όμω ένα ερωτήματα. Αυτά τα εκθέτουμε στην τελογική έκθεση του κειμένου μας. Αφορούν τα ασφαλιστικά της ΟΣΕΚΑ και επίσης τον υπολογισμό των αποδόσεων. Άλλο σημείο που μας ανησυχεί δεν το λέμε στο κείμενο του ψηφίσματος, αλλά Το έχουμε πει με πολλούς συναδελφούς ότι δηλαδή θα πρέπει να αναβληθεί η θέση σε ισχύ του νομοθετήματος. Οπότε και είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή και ο κύριος Μπερναρντίνο να μας διευκρινίσουν τι ισχύει, σε ποιο νομικό πλαίσιο κινούμεθα. Εάν τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία σε πρώτο επίπεδο, τι θα γίνει. Εάν δεν ε, τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα και τα Είμαι εδώ που υπάρχει κάποια σύγχυση ε, και είναι κάπως ασύμμετρη αυτή η ρύθμιση. Οπότε ελπίζουμε να δοθούν απαντήσεις. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Μπάλτς για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο, ο κ. Πιετικάινεν και ο συγητής ε, μου ζήτησε να τον... Η, η, η κυρία Πιετικάινεν κυρία Πιατικά είναι σκιώδη ηγήτρια μου ζήτησε να την αντικαταστήσω ε, σήμερα. Ε, ο στόχος είναι να παρέχουμε διαφάνεια και σαφήνεια ε, μεταξύ των διαφόρων πακέτων δεσμών ε, Διότι αυτά απευθύνονται σε διαφορετικούς τύπους ε, καταναλωτών, πελατών και θα πρέπει αυτοί να έχουν τη δυνατότητα σύγκριση ανεξαρτήτως από πού αγοράζουν αυτά τα προϊόντα. Συνεπώς οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι απλές, ευανάγνωστες και να είναι κατανοητές ακόμα και στους λιγότερο ε, έμπειρους. Οπότε η νομοθεσία θα πρέπει να εξισορροπήσει ε, την, ε, το χειρισμό των διαφόρων προϊόντων. Ε, η η σκιώδηση γήτρια θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της ε, νομοθεσίας δεν αντικατοπτρίζεται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές όπως προτείνονται, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα προϊόντα πολλαπλών επιλογών και του βιομετρικού και πιστοτικού κινδύνου για ε, τέτοιου είδους προϊόντα. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε την Κομισιόν και την ΕΙΟΠΑ. Ε, θα μπορούσαν να μας εξηγήσουν τις ε, επιλογές που έχουν κάνει στον ε, κατεξοδότης κανονισμό. Η ομάδα μας επίσης ε, ανησυχεί και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του κανονισμού. ενδεχομένως θα μπορούσαμε να αναβάλουμε την εφαρμογή του, αλλά με πολύ προσοχή σοφροσύνη θα πρέπει να το εξετάσουμε προσεκτικά. Ε, συνοψίζοντας, η κυρία Πιετικάινεν ε, υπογραμμίζει ότι είμαστε ε, προσιλωμένοι στο περιεχόμενο του κανονισμού και εγώ ίδιος θα ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό. Ευχαριστώ. Um, Ο κύριος Καμάλ, ευχαριστώ. Όλα αυτά τα χρόνια επεξεργαζόμεθα νομοθετικά μέτρα, ακούμε υπέρ και κατά, βγάζουμε κρίσεις σχετικά με το τι πιστεύουμε ως θεμητό και τι απορρίπτουμε ως ιδιωτελές. Εδώ κάποιες ανησυχίες για τα τεχνικά πρότυπα από τον κλάδο, πολλά, ε, πολλές ανησυχίες, κάποιες δεν είναι, κάποιες είναι θεμητές από εταιρείε που είναι συνεργάσιμες γενικά, δεν είναι αντιδραστικές στη νομοθεσία, ενδιαφέρονται για τη φήμη τους και τους καταναλωτές. Λοιπόν, συμφωνώ με πολλά που ακούστηκαν από τον εκπρόσωπο του ΕΛΚ. Ευχαριστώ την Κομισιόν που ήρθε σήμερα. Έχω μια ερώτηση άμεση. Αν απορρίψουμε αυτά τα πρότυπα, τι θα γίνει μετά, πόσο γρήγορα μπορεί να αντιδράσει η Κομισιόν και τι θα κάνει για να μετριάσει θέματα ευθύνης που θα προκύψουν αν δεν υπάρξουν τα RTS, δηλαδή τα αριθμιστικά τεχνικά πρότυπα. Ε, Φιλελεύθερη, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να προσθέσω στους προλαλήσαντες. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα η κατεξουσιοδότηση η πράξη που εγκρίθηκε τον Ιούνιο φοβούμαι ότι δεν είναι σαφής και τα θέματα που δημιουργούν ανησυχία από μας ε, κατεγράφησαν, κάποιοι επαναφέρθηκαν και τώρα. Θα πρέπει να γίνει ό,τι καλύτερο για να διορθωθεί με τρόπο διαφανή η κατάσταση και βέβαια δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε λάθος στα μέτρα του επίπεδου 2. Θέλω επίσης να ακούσω το χρονοδιάγραμμα της Κομισιόν. Αυτό το ζήτησαν και οι προηγούμενοι ομιλητές άλλωστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για την ΚΟΕ. Ο σκιώδης μας λείπει, οπότε αν θέλετε μπορείτε να συνεχίσετε με τους υπόλοιπους σκιώδης ηγητές και μεταξύ θα επιστρέψει. Okay. Sven Giegold. Καλώς, Sven Giegold. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να τονίσω για λογαριασμό της ομάδας μου ότι είμαστε υπέρ του στόχου των πρίψε να γίνεται καλή ενημέρωση των καταναλωτών και να αυξάνεται η συγκρισιμότητα των προϊόντων για τους τελικούς καταναλωτές για να ανοίξει και η αγορά των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Υπάρχουν τμήματα του κλάδου που δεν το θέλουν αυτό γιατί οι πρόσοδοι τους θα μειωθούν και ξέρουμε ότι υπήρξαν πολλές πιέσεις κατά τις διαπραγματεύσεις ε, του κειμένου επίπεδου 1 ήδη. Δεν είμαστε απλοϊκοί. Δεν θεωρούμε ότι οι ενστάσεις αυτές ε, θα εξυπηρετήσουν ανθρώπους που δεν θέλουμε. Κατόπιν τούτου, νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το κείμενο του επίπεδου 1 δεν ε, είναι όριμο για διαπραγματεύσεις εμείς θέλουμε να εφαρμόσουμε την νομοθεσία, αλλά σωστά, με τρόπο μη παραπλανητικό. Και εδώ πρέπει να πω ότι δεν είμαι καθόλου ευτυχής με την ε, λειτουργία της συνεργασίας. Εμείς δώσαμε στην Κομισιόν και στην ΕΣΜΑ ε, πολύ νωρίς ε, τα, τις ανησυχίες μας και είπαμε ότι τα δεδομένα που παρουσιάζονται με τρόπο γραφημάτων ε, είναι παραπλανητικά για τους καταναλωτές. Εμείς δώσαμε υπολογισμούς για πολλά ταμεία ε, και τίτλων και εκείνη της περιουσίας, ε, αξιογράφων και εκείνη της περιουσίας και αν δούμε προηγούμενα στοιχεία και θεωρήσουμε ότι η πρίψη ίσχυε από τότε και αν κάνουμε προβολή στην επόμενη πενταετία Βλέπουμε ότι αν ήταν δυσμενή τα σενάρια μετά, τα στοιχεία θα ήταν ή πολύ, ε, θετικά ή πολύ αρνητικά στο 1 τρίτο των περιπτώσεων σε περίπτωση αγοράς και η αξία της επένδυσης θα μειωνόταν αλλά ακόμα και στο δυσμενές αλλά θα μειωνόταν η, επένδυ, η αξία της επένδυσης αλλά ακόμα και το χειρότερο σενάριο θα άδειχνε κέρδη. Αυτό είναι πολύ παραπλανητικό. Εμείς ε, θέλουμε ε, να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι η νομοθεσία αρχίζει να ισχύει σε περίοδο χαμηλών επιτοκίων. Ε, έτσι λοιπόν θα πρέπει, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι θα χρειαστούν διορθώσεις. Αν τώρα δώσουμε ε, πληροφορίες λάθος, επειδή οι προηγούμενες πληροφορίες έπαιξαν ρόλο ε, σημαντικό για τα σενάρια θα δώσουμε λάθος πληροφορίες ότι και στο δυσμενές σενάριο είναι πιθανόν να έχουν κέρδη όταν επενδύσουν ε, σε ακίνητα ή στις μετοχές ή οτιδήποτε σε κινητές αξίες. Και τότε θα έρθουν, θα να μας χτυπήσουν την πόρτα σε εμά τους ευρωβουλευτές και θα μας θεωρήσουν υπεύθυνου. Θα πούνε εγώ έχασα στο χρηματιστήριο λεφτά, ενώ η ενημέρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έδειξε ότι υπό δυσμενείς συνθήκες υπάρχει κίνδυνος από ζημιάς. Ε, το λέω και στους ε, φιλελευθέρους φίλους. Δεν θέλω να αποτρέψω τον κόσμο από την ανάληψη κινδύνου. Πολλοί άνθρωποι έχουν μόνο ε, καταθετικούς λογαριασμούς και, από σε τα... Ε, και Ε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάσουν και λεφτά και εδώ παραπλα... είναι παραπλανητικές οι πληροφορίες. Ενημερώσαμε την Κομισιόν, ενημερώσαμε και την ΕΣΜΑ την αρχή αξιών και αγορών. Ε, είπαμε να τσεκάρουν τα στοιχεία και να δουν αν είναι σωστά. Μέχρι τώρα κανείς δεν μας απάντησε να μας πει αν επιβεβαιώνουν την ορθότητα των στοιχείων. Ε, έγιναν κάποιες συζητήσεις και ευχαριστώ τους υπεύθυνους στη Κομισιόν και στην ΕΣΜΑ που έκαναν αυτές τις συζητήσεις για να δούμε πώς θα λυθεί το πρόβλημα, αλλά ακόμα λύση δεν έχουμε βρει. Και τώρα θα πρέπει να διορθώσουμε την κατάσταση, γιατί στο επίπεδο 1 λέει η νομοθεσία ότι δεν μπορεί να είναι τα στοιχεία παραπλανητικά. Και ένα δεύτερο που μας ενοχλεί είναι ότι στις διαπραγματεύσεις ε, ως κοινοβούλιο είχαμε το Comprehension Alert, όταν δηλαδή είναι υπερβολικά περίπλοκα τα προϊόντα. Υπάρχει ένα σήμα κινδύνου. Αλλά στο RTS, τα τεχνικά πρότυπα, δεν υπάρχει τώρα ε, κάποια ενημέρωση ε, για το, τα σήματα αυτά. Οπότε η ΕΟΠΑ να μας πει, μπορείτε να μας το διευκρινίσετε, ότι δηλαδή αυτό το σήμα κατανόησης, το Comprehension Alert, θα χρησιμοποιείται με νέο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί με την ε, Ένωση ε, Κεφαλαίου Αγορών θέλουμε ισότιμους κανόνες παντού για να μπορεί να λειτουργήσει η ε, Ένωση, Κεφαλαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, ναι στα, στους στόχους του, του ΠΡΙΠΣ, αλλά θέλουμε η Κομισιόν και οι εποπτικές αρχές να συνεργάζονται καλύτερα όταν τίθενται τέτοια σοβαρά ζητήματα. Ευχαριστώ. Άλλους ομιλητές δεν βλέπω. Ο Τζον Μπάριγκαν από την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε αυτή την σημαντικότατη συζήτηση. Ο κανονισμός ΠΡΙΠΣ και οι σχετικές ε, διατάξεις για τις ε, βασικές πληροφορίες είναι σημαντικό βήμα για να βελτιώσουμε την διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο. Ιδιαίτερα το αναφορεί τις βασικές πληροφορίες για πρώτη φορά θα εισάγει κοινά προδιαγραφές για το πώς θα παρουσιάζονται οι πληροφορίες σε μια ευρεία γκάμα επενδυτικών προϊόντων. Αυτό θα βοηθήσει τους επενδυτές να μπορούν να συγκρίνουν ε, τις, ε, τα χαρακτηριστικά, το κόστος και την μελλοντική απόδοση αυτών των προϊόντων και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να πάρουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. Ας το έχουμε υπόψη μας αυτό λοιπόν στη συζήτηση. Στις 30 Ιουνίου το Κολέγιο των Επιτρόπων ενέκρινε αυτόν τον ε, κατεξιόδοτη κανονισμό ε, που περιλαμβάνει τι λεπτομέρειες για το, και τεχνικές προδιάρφες για την παρουσίαση των πληροφοριών. Ε, ο χρόνος μας πίεσε πάρα πολύ στην ε, προετοιμασία του κανονισμού. Παρ' όλα αυτά, Κάναμε χρήση των ε, συμβουλών της ομάδας συμπρογνωμόνων, ε, μια ευρεία ε, διαβούλευση και μια ακρόαση. Με βάση όλα αυτά καθορίσαμε τις ψηλές αυτές, ψηλών απαιτήσεων προδιαγραφές που είναι υπέρ των συμφωνών των καταναλωτών. Ο Γκάμπριελ θα σας εξηγήσει με περισσότερες λεπτομέρειες αυτές μας επιλογές. Το περιεχόμενο όμως ε, του κανονισμού ε, ε, βασίζεται και στη δική μας εμπειρία. Είμαστε σίγουροι ότι τα προτινόμενα καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών. Η Κομισιόν επίσης πολύ γρήγορα υιοθέτησε τον ε, κατεξόδοτης κανονισμό. Όπως είπε ο Πρόεδρος κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του κανονισμού ε, σας κρατήσαμε ενήμερους και για την ουσία αλλά και για το χρονοδιάγραμμά μας. Αντιλαμβάνομαι πως υπάρχουν κάποια θέματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και σε σχέση ιδιαίτερα με την επιστολή της ΕΚΟΝ που έφτασε τέλος Ιουνίου μετά την υιοθέτηση του κανονισμού. Λυπηρό, αλλά να είμαι σαφής. Ε, δεν αποτελεί έλψη σεβασμού από δικαίωνος πλευράς. Ο λόγος για τον οποίο υιοθετήσαμε αυτόν τον κανονισμό τόσο γρήγορα ήταν η προθεσμία που είχαμε. Θέλαμε να δώσουμε στον κλάδο ε, αρκετό χρόνο για να προσαρμοστεί. Αναγνωρίζουμε ότι η προθεσμία για τον κλάδο είναι, εξακολουθεί να είναι πολύ στενή, οπότε κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την εφαρμογή. Ένα workshop ε, που διοργανώθηκε τον Ιούλιο ήταν ένα από τα μέτρα, μία από τις δράσεις μας και είμαστε έτοιμοι ε, να εκδώσουμε ε, εγχειρίδιο και για το επίπεδο 1 και για το επίπεδο 2. Προσπαθούμε λοιπόν να βοηθήσουμε τον κλάδο να προσαρμοστεί μέχρι την προθεσμία. Η Κομισιόν μαζί με τις εποπτικές αρχές μετά την εφαρμογή θα ε, εξετάσει το πώς εφαρμόζεται ο κανονισμός και αυτό θα μας επιτρέψει να, βρούμε που χρειάζεται, να δούμε πού χρειάζεται περισσότερη δράση για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε προβλήματα εμφανιστούν. Το πλαίσιο PRIMS είναι ένα πρώτο βήμα για να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη διαφάνεια των επενδυτικών προϊόντων. Για μας είναι σημαντικό όμως βήμα. Ε, το, ε, η, η ρυθμιστική τεχνική προδιαγραφή αποτελεί ε, ένα συμβασμό μεταξύ των συμφερόντων όλων. Οπότε όλοι τέτοιου τύπου συμβιβασμοί προφανώς δεν ικανοποιούν 100% τους πάντες. Πρόκειται για συμβιβασμό. Πιστεύουμε όμως ότι οι μικροεπενδυτές θα ε, ωφεληθούν ιδιαίτερα. Ε, θέλουμε να μέχρι το τέλος της προθεσμίας, δηλαδή το τέλος του χρόνου, να είναι σε ισχύ όλο το πλαίσιο PRIMS. Ε, η καλύτερη βέβαια λίστα ήταν και ο κανονισμός και PRIMS και ο κατεξοδότης κανονισμός να εφαρμοστούν ταυτόχρονα. Η, η εξέταση αυτή τη τεχνική προδιαγραφή θα οδηγούσε όμω ε, σε ε, καθυστέρηση στην εφαρμογή και του σχεδίου κανονισμού. Οπότε, αν θέλετε να απορρίψετε τον κατεξοδότη κανονισμό, εμεί θα συνεχίσουμε να συνεργαστούμε μαζί σα για ένα συμβιβασμό που θα ικανοποιεί τι ανησυχίε όλων, έτσι ώστε η τεχνική προδιαγραφή να μπει σε ισχύ το συντομότερο δυνατό και έγκαιρα έτσι ώστε να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα όλων. Παρ' όλα αυτά, με βάση της, ε, ε, τη γνώμη της νομικής μας υπηρεσίας, της νομικής μας ε, ο, ο, το επίπεδο 1 εξακολουθεί να ισχύει και υπάρχουν ε, στον κανονισμό διατάξεις που, αρχίζουν να ισχύουν από τις 31 Δεκεμβρίου του 2016 οπότε ε, ο, κανονισμό κανονισμός επίπεδου 1 δίνει αρκετέ πληροφορίε στον κλάδο, έτσι ώστε να προχωρήσει ακόμα και χωρί τον κατεξοδότη κανονισμό. Η δεύτερη, βέβαια, λύση δεν θα ήταν η καλύτερη. Θα δημιουργήσει μια, ένα νομικό κενό και θα αύξανε το κόστος. Ε, ο καθένας θα δημιουργούσε τις δικές του ε, μεθοδολογίες ε, για την παρουσίαση των στοιχείων με βάση τα όσα λέει ο κανονισμός. Ε, και μετά την υιοθέτηση του, της καινούργια RTS θα πρέπει να προσαρμόσουν αυτά που είχαν αποφασίσει. Η Κομισιόν θα προσπαθήσει να μετριάσει τα προβλήματα ε, και να μειώσει τον κίνδυνο μη συγκρισιμότητας, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό θα το καταφέρουμε έγκαιρα. Δεν είναι η καλύτερη λύση αυτή. Παρόλα αυτά, ακόμα και αυτή η λύση αποτελεί σημαντική βελτίωση της σημερινής κατάστασης. Συνοψίζοντας, ο κατεξοδότης κανονισμός πιστεύουμε ότι όπως εγκρίθηκε από την Κομισιόν είναι ο καλύτερος τρόπος για την εφαρμογή ε, του ε, κανονισμού. Αν απορριφθεί, ο κανονισμός πρέπει θα εξακολουθήσει και πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται. Δεν είναι η καλύτερη λύση. Παρόλα αυτά, είναι καλύτερο από το να μην έχουμε κανένα νομοθετικό κείμενο. Για να αποφύγουμε σε αυτή τη δεύτερη λύση, μπορούμε να συνεχίσουμε, είμαστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε να συνεργαστώ μαζί σας για ένα συμβιβασμό που θα μας επιτρέψει να αρχίσουν να, να τεθούν σε ισχύ και τα δύο κείμενα, και ο κανονισμός και ο κατεξουδότης κανονισμός ταυτόχρονα. Ευχαριστώ. Thank you. I have to say a bit of calling this second scenario. Ευχαριστώ. Το δεύτερο το λέτε δεύτερο σε προτίμηση, προτιμητέο δηλαδή ως δεύτερο. Με έκπληξη το άκουσα αυτό. Ο κύριος Μπερναρντίνο, ευχαριστώ. Καταρχήν, ε, ευχαριστώ που βρίσκομαι εδώ αφού μας δώσατε ευκαιρία να συζητήσουμε το σημαντικό έργο αυτό, τα ρυθμιστικά τεχνικά πρώτη RTS για τα πρίψ που είναι σημαντικά για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Το σχέδιο αντικατοπτρίζει πολλά έτη δουλειάς από τα μέλη των τριών εποπτικών αρχών. Πολλές προσπάθειες έγιναν για να βρεθεί δίκαιη προσέγγιση για όλα τα πρίψε. Ε, και τους κατασκευάστες, τους προμηθευτές τους. Έγιναν πολλές διαβουλεύσεις, ε, τρεις χωριστές ε, και υπήρχε και ομάδα εμπειρογνωμόνων. Επίσης ακούστηκαν και οι γνώμες των καταναλωτών. Από νωρίς είδαμε ότι έπρεπε να βρεθεί ισορροπημένη λύση, συμβιβαστική, και τα μέλη των ρυθμιστικών αρχών κατέληξαν σε αυτά τα RTS. Τώρα να δούμε το κόστος και ποιο είναι για τα διάφορα πρίψ. Πιστεύουμε ότι το πακέτο βελτιώνει πολύ τη διαφάνεια και συγκρισιμότητα του κόστους. Θέλω να τονίσω εδώ ότι ρητά δεν θεωρούμε κόστος το βιομητρικό ασφάλιστρο κινδύνου, αλλά βάζουμε στο κόστος μόνο το κομμάτι του ε, βιομετρικού ασφάλιστρου κινδύνου που είναι 100% κόστος. Και αυτό είναι δίκαιο. Δουλέψαμε σκληρά για να βρούμε παρόμοια ισορροπία δίκαιη και για τους κινδύνους. Ε, τώρα για τον πιστοτικό κίνδυνο πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να, να, να τον αναγνωρίσουμε όποτε προκύπτει και αυτό μπορεί να ε, συμπεριλαμβάνει ασφαλιστές που υπόκεινται στο Solvency 2. Να είναι ξεκάθαρο αυτό, γι' αυτό δεν έχουμε γενική απαλλαγή των ασφαλιστών. Ε, στο σχέδιο RTS πιστεύουμε ότι γίνεται καλή προσπάθεια εξέβρεσης λύσης αναγνωρίζομαι και ρόλο πληρεξούσιου αλλά και ε, ε περιπτώσεις μετριασμού του πιστοτικού κινδύνου ε, όπως ε, υπάρχει, όπως είναι δεδομένο για τους ασφαλιστές, τους περισσότερους ε, υπό Solvency 2 πρέπει να ε, γίνουν μεταρρυθμίσεις βέβαια στα πλαίσια του Solvency 2 που θα διευκολύνουν και άλλες λύσεις και θα αποκαταστήσουν μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτό αναφέρεται και στο σημείο 6 του ε, σχεδίου του RTS. Για να δούμε τώρα το ε, σενάριο της απόδοσης. Καταλαβαίνουμε βέβαια και είναι αλήθεια ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί λύση ε, βάσει, διαφορετικών, ε, βάσει προηγούμενης ε, απόδοσης να δούμε τα σενάρια. θα πρέπει να δούμε καλύτερα τα δυσμενή σενάρια. Δουλέψαμε πάνω στην πιθανή χρήση που προβλέπεται στο σχέδιο RTS του πρώτου σεναρίου για να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις καταστάσεις όπου το α δυσμενές σενάριο μπορεί να φαίνεται υπερβολικά ρόδινο κάποιες φορές, αλλά πιστεύομαι ότι αυτό που έχουμε στο σχέδιο RTS θα είναι αρκετό για να έχουμε πρακτική εφαρμογή του, η οποία θα έλεγα θα εξασφάλιζε όχι παραπλανητική εικόνα, αλλά δίκαιη εικόνα στους καταναλωτές. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι έχουμε κάποια κατανόηση σε επίπεδο των ε, ρυθμιστικών αρχών ε, εις ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του πακέτου. Δεν είναι καινούριο αυτό, το έχω ξαναπεί την περασμένη φορά που ήρθα για να το συζητήσουμε αυτό. Σκεφτήκαμε ότι έπρεπε να είναι βέβαιο ότι θα περάσουν στην εφαρμογή τα σχέδια αρτίες. Όπως είπαμε και τότε, γνωρίζαμε τις προκλήσεις ε, του κλάδου λόγω του μικρού χρονοδιαγράμματος στενού. Δουλέψαμε για να ε, έχουμε ερωταπαντήσεις ε, και άλλα, άλλο υλικό για να πάρουμε στοιχεία από τον κλάδο. Και όπως είναι φυσιολογικό, τα μέλη των ρυθμιστικών αρχών συζήτησαν ευρύτατα με τους, όλους τους εμπλεκομένους θέματα εφαρμογής. Ε, θέλουμε και έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν καλά στον κλάδο και ε, τα, τα ε, πρότυπα αυτά. πρέπει όμως να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι ρεαλιστική η προσέγγιση στο νέο καθεστώς. Τέλος, το θέμα του Comprehension Alert, ε, σήμα κινδύνου. αυτό δεν ήταν κομμάτι της εντολής που μας ανέθεσε η Κομισιόν και νομίζω ότι ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Δεν ήταν αυτό τμήμα του προτύπου, πάντως ε, είμαστε έτοιμοι να το δούμε και αυτό αν μας αναθέσει η εντολή η Κομισιόν να ασχοληθούμε με την πρακτική εφαρμογή του Comprehension Alert. Ευχαρίστως θα είμαστε ευτυχείς να ανταποκριθούμε. Τώρα, κοιτάζοντας το μέλλον και καταλαβαίνουμε βέβαια τις ανησυχίες σας, είμαστε έτοιμοι ε, οι ρυθμιστικέ αρχέ ε, να δουλέψουμε και με την Κομισιόν και με τον Κοινοβούλιο για να διευκρινίσουμε και να βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουμε ε, όπω πρέπει τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν. Πρέπει να πω ότι στη δουλειά που κάναμε στις ερωταπαντήσεις για την εφαρμογή του σχεδίου των RTS ε, παρουσιάσαμε και πρακτικές λύσεις. Κάποιες από αυτές σίγουρα ε, προσεγγίζουν τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου σε πολλούς τομείς. Πιστεύω και είμαι αισιόδοξο ότι αν όλοι συνεργαστούμε με πνεύμα κατάλληλο, δηλαδή να υπηρετήσουμε τους καταναλωτές, ε, αυτό είναι το καθήκον όλων μας, μπορούμε να τα ε, θέσουμε σε εφαρμογή όλα αυτά με ωραίο και έγκαιρο τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Κύριε Περνέντο και κύριε είναι σημαντικό, νομίζω, όσα μας εξήγησε ο κύριος Μπέργαν. Πρόκειται περί συμβασμού. Πολιτικοί είμαστε. Ξέρουμε ότι πρέπει να συμβαζόμαστε. Δεν ξέρω τώρα, ε, εκεί είναι το θέμα το κατά πόσο είναι συμβασμός. Ο συμβασμό είναι συμβασμό, αυτό αφορά και το κοινοβούλιο. Αλλά, αλλά κινείστε στα πλαίσια του συμβασμού. Οπότε, είμαι λίγο στριμωγμένος. Πώς θα τα συγκεράσουμε αυτά, το περιεχόμενο, την ουσία, με τον συμβιβασμό. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι. Έχουμε εδώ συγκεκριμένα προβλήματα. Και τι θα κάνουμε τώρα στο βωμό του συμβιβασμού. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε για κάποια έγγραφα τα οποία δεν βοηθούν στο να συγκρίνει κανείς τα προϊόντα. Μα ο συμβιβασμός δεν είναι αυτός ο σκοπός. Θα πρέπει να ωφελεί σε κάτι. ξέρω εάν αυτά τα επιχειρήματα είναι πιστικά, εάν καλύπτουν τα πολύ συγκεκριμένα προβλήματα που αναδείχθηκαν. Οπότε νομίζω τώρα απόκειται στους βουλευτές να μας πούνε αν επί της ουσίας καλύπτονται ή όχι. Σας επαναλαμβάνω. Η πρώτη μου αντίδραση είναι έκπληξη που νιώθω. τι θα γίνει με την κατεξοδότηση πράξη. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουν οι βουλευτές. Περβάμψω. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Μπερναρτίνο και τον συνάδελφο από την Κομισιόν για την ε, παρουσιάση του και τις απαντήσεις τους. Ε, ασφαλώς η, πρέπει να σχολιάσουμε το θέμα της θέσης ισχύω του κανονισμού χωρίς την, ε, το RTS, χωρίς τον κατεξίοδο της κανονισμού. Ε, υπάρχει βέβαια μια ανησυχία για το κατά πόσο θα γίνει ομοιόμορφη εφαρμογή. Αλλά το ερώτημα είναι το εξή. Ε, στην επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος της Επιτροπής ΕΚΟΝ στον Επίτροπο, σε ποιο σημείο η Κομισιόν και η ΟΠΑ είναι πρόθυμες να διαπραγματευτούν για να βελτιωθεί η κατάσταση. Πρέπει να ξέρουμε, δηλαδή, τι προοπτικές υπάρχουν για την βελτίωση του κατεξουδότης κανονισμού. Ο κ. Μπάλτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Τζον ε, Άρεγκαν και τον Γκάβριλ Μπερναντίνον για τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων. Ε, Εμεί ως Επιτροπή ΕΚΟΝ στα... έχουμε επιφυλάξει για τα τεχνικά πρότυπα αυτό το έμαθε η Κομισιόν ε, έγκαιρα. Θέλαμε λοιπόν πριν από την έγκριση της νομικής πράξης να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πιο συγκεκριμένες προσαρμογές και τροποποιήσεις στα σχέδια. Βεβαίως ε, η Κομισιόν έχει το προνόμιο, δεν το αμφισβητεί κανείς, να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξης. Αλλά και το Κοινοβούλιο έχει το προνόμιο να απορρίπτει τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις αυτές και Θέλω να το πω καθαρά, εξ ονόματος ολόκληρης της ομάδας μου, του ΕΛΚ, ότι σε σχέση με την διοργανική συνεργασία ε, θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερους συσχετισμούς. Είναι σαφές για την ομάδα μας ότι μια δήλωση σε επίπεδο κατεξουσιοδότηση πράξεων είναι χρήσιμη. Εκεί όπου υπάρχουν διαφορές θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε το θέμα ε, με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Αν ε, δεν συμμετέχει το Κοινοβούλιο, αυτό θα το θεωρήσουμε απαράδεκτο. Επίσης, η ασφάλεια δικαίου για τους καταναλωτές είναι ε, ζητούμενο, γιατί αυτοί σε τελευταία ανάλυση θα αξιοποιήσουν τα έγγραφα αυτά, τα έγγραφα βασικών πληροφοριών. Ξέρουμε ότι μια τροποποίηση στις κατεξουσιοδότηση πράξης έχει συνέπειες και για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των πρίψε Όμως, να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα από την πλευρά μου. Δεν θέλω να αναβληθούν επάπειρον τα πρίψε, γιατί και προσωπικά έχω τα... θεωρώ ότι ε, η ενημέρωση, αν ενισχυθεί ε, και αν ε, παρέχεται με ενιαίο τρόπο προς τους καταναλωτές, αυτό είναι ζητούμενο και γι' αυτό χρειάζεται ο κανονισμός πρίψε και οι σχετικές ε, κατεξουσιοδότηση και η σχετική κατεξουσιοδότηση πράξη. Και μάλιστα, όπως είπε και ο Τζον Μπάριγκαν, θα πρέπει ταυτόχρονα να δεθούν σε εφαρμογή όλα αυτά. Πρέπει να δούμε λοιπόν την κατεξουσιοδότηση πράξη και τον κατεξουσιοδότηση κανονισμό, ε, να τα δούμε σε ένα σύνολο. Το second best, η δεύτερη καλύτερη επιλογή, που αναφέρθηκε εδώ δεν νομίζω ότι είναι πρακτική, δεν ε, είναι εφαρμοστέα. Και αναφέρθηκε ο second best, best. Ε, το, το, η λέξη best εδώ δεν αρμόζει, η βέλτιστη δηλαδή, δεν πρόκειται για βέλτιστη. Άρα, η Κομισιόν πρέπει να ξανασκεφτεί τη θέση της. Έχω την εντύπωση ότι όλους μας ενδιαφέρει μια καλή λύση. Ε, θα κάνουμε την ψηφοφορία και θα δηλώσω για την ομάδα μου ότι μετά θα είμαστε αμέσως έτοιμοι για να κάνουμε συζητήσεις με την Κομισιόν, με όλους τους εμπλεκομένους και προφανώς και με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Κύριος Καμάλ. Να σχολιάσω αυτά που είπαν οι Περβάνος και ο Μπέρχαρτ. Θα ήταν καλύτερο βέβαια να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα τα δύο κείμενα. Να ρωτήσω και την Κομισιόν. Ε, αυτό που ρώτησε η κυρία σε ποια σημεία είναι πρόθυμη η Κομισιόν να διαπραγματευτεί. Ε, επίσης, με προβληματίζει η Κομισιόν να θέλει το περιθώριο να αγνοήσει μια απόρριψη, μια έκφραση αντιρρήσεων, οτιδήποτε και να γίνει δηλαδή. Ε, δεν θα ήθελα, δεν θα μ' άρεσε η Κομισιόν να δείξει ότι αγνοεί την αντιρρήσή μας. Ε, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω. το οργανισμό το ψηφίσαμε και θα τεθεί σε λειτουργία. Αυτό στο οποίο έχουμε αντιρρήσει είναι οι πληροφορίε οι οποίε θα στέλνονται στου καταναλωτέ. Και μερικές ε, φορές οι προδιαρθές ε, οι οποίες θα συμφωνηθούν μπορεί να παραπλανούν τον καταναλωστή. Ε, ε ασφαλώς και συνήθως λέμε ότι μπορεί η απόδοση να είναι θετική και, αλλά και αρνητική, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Αντιπαθώ τέτοιου είδους ε, φράσεις. Το καλύτερο είναι να λέμε να επενδύσετε χρήματα μόνο όταν είστε διατεθειμένοι να τα χάσετε, όταν είστε έτοιμοι να τα χάσετε κιόλας. Αυτό θα πρέπει να λέμε στον καταναλωτή. Κύριος Γιάζεκ. You don't have to, but... Δεν χρειάζεται να πάρει το λόγο. Ο Κύριε um, um, Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, νομίζω ότι σήμερα σημειώθηκε μια κάποια πρόοδος και είναι σαφές ότι υπάρχουν δύο απόψεις γιατί θα πρέπει να απορριφθεί αυτή η κατεξουδότηση πράξη. Τα λέμε ξεκάθαρα. Οι περισσότεροι θέλουμε να τεθούν οι κανονισμοί ταυτόχρονα σε ισχύ και μέσα στο πλαίσιο που έχει καθοριστεί. Ο Σβήν μας πει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και αυτά τα θέματα θα πρέπει να αναφερθούν στις ε, επαφές μας με την Επιτροπή. Η Επιτροπή εδώ και μήνες λέει τα ίδια αλλά και ο Σβέν το ίδιο προς τιμήν του. Και θα πρέπει να ισχύσει το σενάριο που προτιμώ εγώ, δηλαδή το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Όσο γίνεται. Και έχουμε μετά βέβαια και το δεύτερο καλύτερο, αυτό που μας λέει η Επιτροπή. Όμως, Δεν ξέρω πώ ε, αυτού του είδου η αντιμετώπιση αντικόκτηση μπορεί να αποκαταστήσει την αρχική ρύθμιση για τα αρτίες. Με τι χρονοδιάγραμμα θα λύσουν τα θέματα αυτά, πώς θα τα θέσουν όλα αυτά σε εφαρμογή στο πλαίσιο που αρχικά είχε αποφασιστεί. Ευχαριστώ. Σβέν. Πρώτα πρώτα. Ευχαριστούμε για την ε, προθυμία σας να συνεχίσουμε την ε, αναζήτηση κάποιες λύσεις. Και σας τονίζω. Σίγουρα δεν βοηθάει το ότι αυτά τα δύο σημεία τα οποία εμείς προσθέσαμε στην αρχή σας πρόταση δηλαδή τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα και το comprehension alert Αυτά τα δύο. Τα πρότεινε το κοινοβούλιο. Και πού πήγαν αυτά. Ξεχάστηκαν. Ενώ η Κομισιόν ήταν υποχρεωμένη αυτά να καλυφθούν στο δεύτερο επίπεδο δεν έγινε τίποτα. Αυτά ξεκίνησαν πριν καν. Πάρετε κύριε το, το αξίωμα, τη θέση που έχετε τώρα το Comprehension Alert και η άλλη ρυθμίση που προτείναμε. Να μας παίρνετε στα σοβαρά. Έτσι να προχωρεί η δουλειά σας. Εμείς παίρνουμε σοβαρά τη δική μας δουλειά. Και έτσι όπως τα πάτε θα έχουμε πρόβλημα. Τα έρθει η εδώ. Εμείς πάντοτε είμαστε φιλοευρωπαίοι, ε, θέλουμε να καλύψουμε τον καταναλωτή, φυσικά και μας καίει το νομοθέτημα. Αυτό είναι το μήνυμα που σας στέλνουμε, κύριε Μπερναρντίνο. Πώς θα λύσετε αυτό το πρόβλημα εδώ, βλέπετε τι λέει αυτό το γράφημα, αυτή η γραφική παράσταση. Όσο πιο γρήγορα προχωρήσετε τόσο καλύτερα, αλλά να είναι αξιόπιστη η λύση. Έτσι δεν έχουμε καμιά οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Έχετε το κείμενό μας στο σχέδιο του ψηφίσματος. Δεν μας έχετε καλύψει, δεν απαντήσατε σε τίποτα. Το είπα και στον κύριο Γιέζεκ. Αυτό κάπως θυμίζει τις κεντρικές επιτροπές απαντάνε χωρίς να πάνε επί της ουσίας. Και λένε, α, ωραίος, ισόρροπος, συμβασμός κλπ. κλπ. Εμείς είμαστε περήφανοι που γκρεμίσαμε το, την Κεντρική Επιτροπή των Κομμουνισμών. Τι να τα κάνουμε όλα αυτά τα στρογγυλά και όλα τα δίθεν στοιχεία, γιατί άλλα λένε τα πραγματικά στοιχεία. Πολλέ φορέ φαίνονται όλα στο κοιλάκι ότι θα προκύψουν κέρδη, ενώ τελικά το αποτέλεσμα είναι μόνο ζημία. Οπότε, για κοιτάξτε τα καλά, φέρτε μα κάποια ουσιαστική λύση, οπότε και εμεί τότε θα είμαστε ανοιχτοί για να μπορέσουμε να βρούμε ε, κάποια, κάποια, τέτοια, κάποια λύση. Αλλά μην, μας, ε, μην ακολουθείτε τη μέθοδο τη Κεντρική Επιτροπή, γιατί είδατε τι έγινε δεκαετία του 90. Πρόεδρος, Μπέργεν και Μπερναρντίνο. να απαντήσω ορισμένα από τα σχόλια που έγιναν. Ε, όχι με χρονολογική σειρά, αλλά με σειρά σημασία ενδεχομένω. Η Κομισιόν προτιμά όλο το νομοθετικό πλαίσιο PRIMS να ε, είναι σε ισχύ πριν τη λήξη προθεσμίας. Ας μην γίνει καμία παρανόηση. Μέχρι το τέλος του χρόνου θέλουμε όλο το πλαίσιο να τεθεί σε λειτουργία προς όφελος των καταναλωτών. Στο, στην, στον κανονισμό όμως, στο, στην νομοθετικό κείμενο επέδου ε, υπήρχε συγκεκριμένη προθεσμία που δεσμεύει τον κλάδο και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την σεβαστούμε. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες. Η εντολή έχει ήδη σταλεί, κύριε Γκίγκολ. Δεν ήταν θέμα προτεραιότητας. Η δεύτερη καλύτερη λύση. Είμαι οικονομολόγος, ε, ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιήσει άλλο, ε, όρο. Σίγουρα η δεύτερη λύση είναι πολύ χειρότερη από την πρώτη, αλλά σίγουρα είναι καλύτερο από το να μην έχουμε τίποτα. Ιδιαίτερα δεδομένη της προθεσμίας την οποία έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω του νομοθετικού κειμένου. Ζητώ συγγνώμη αν η ορολογία που χρησιμοποίησα σας μπέρδεψε. Θεωρώ ότι απλώς η δεύτερη λύση είναι καλύτερη από το να μην έχουμε τίποτα. Ε, μπορούμε να αποφύγουμε πλήρως ε, τις ασυμβατότητες. Ε, όχι. Ε, μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μετριάσουμε το πρόβλημα απλώ Σε αυτή τη δεύτερη καλύτερη λύση, στη, στη χειρότερη από τις δύο λύσεις δηλαδή για το χρονοδιάγραμμα. Ο Γκαμπριέλ ε, είπε ότι συμφωνεί με το χρονοδιάγραμμα και εμείς δεν θα έλεγα ότι διαφωνούμε. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να εργαστούμε το, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ε, θέση μας δεν είναι να αναβληθεί η θέση σε λειτουργία. Και επιμένουμε σε αυτό. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον κλάδο να προσαρμοστεί, αλλά δεν είμαστε υπέρ της αναβολής. Επίσης, δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης των θεσμικών διαδικασιών. Γνωρίζουμε τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τους κατε, κανονισμούς. Και θα συνεργαστούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε ακόμα και αν απορρίψετε το κείμενο σήμερα, και εγώ και ο Γκαβριέλ θα συνεργαστούμε μαζί σας για να αναζητήσουμε ε, ρεαλιστικούς συμβιβασμούς στα θέματα που σας ε, ενοχλούν. Ε, δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες για το πώς θα διαπραγματευτούμε. Θα πρέπει να μιλήσω με τον Αντιπρόεδρο, αλλά μπορούμε να εργαστούμε για το θέμα του πιστοτικού κινδύνου, για τα σενάρια, για πολλά θέματα στα οποία μπορούμε να βρούμε συμβιβασμό. Και ένα τελευταίο σχόλιο για το συμβασμό. Όταν μιλώ για συμβιβασμό δεν εννοώ πολιτικό συμβασμό, εννοώ τεχνικό συμβασμό. Προφανώς ε, ο καθένας θα ήθελε ο συμβασμός να λειτουργεί καλύτερα για τον εαυτό του και χειρότερα για τους υπόλοιπους. Αλλά ο τεχνικός συμβασμός θα είναι αποδεκτός, είναι αποδεκτός ε, σε από πλευρά ποιότητα. Θα λειτουργήσει. Είναι λειτουργικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Μπερναρντίνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα να πω δύο πράγματα. Καταρχήν την εφαρμογή του κανονισμού και τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, τα Δεν θα συζητήσω τα νομικά θέματα, αλλά πιστεύω ότι όλοι πρέπει να συνεργαστούμε για να αποφύγουμε άσκοπη ε, έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Γιατί η εφαρμογή χωρίς αρτιές πιστεύω ότι θα δημιουργήσει μεγάλη αβεβαιότητα, πολλά προβλήματα και για τις εποπτικές αρχές που δεν θα έχουν ε, ανταποκριθεί στην εντολή τους, που είναι η συνεπής εφαρμογή της νομοθεσίας. Είναι δύσκολο να έχουμε συνεπή νομοθεσία σε πολλού τομεί όπου έχουμε κατευθυντηρίε γραμμέ, νομοθεσία επίπεδου 2. Αν δεν τα έχουμε και έχουμε μόνο βασικέ αρχέ, είναι δύσκολο να υπάρχει συνέπεια και συνοχή στην ε, ενιαία αγορά. Προτιμώ λοιπόν να συνεργαστούμε από πριν για να αποφύγουμε προβλήματα ασφάλειας δικαίου δεύτερο θέμα που αναφέρθηκε και είμαστε βέβαιοι βέβαια, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στην εξέβρεση λύσεων. Όπως είπα σε πολλούς τομείς που αναφέρθηκαν στις ανησυχίες του Κοινοβουλίου, ε, δουλεύουμε για να λύσουμε το θέμα με βάση ερωταπαντήσεις Είμαι πεπισμένος ότι πολλά στοιχεία από τις ερωταπαντήσεις και τις γνώμες μπορούν να ενσωματωθούν στα αρτιές για να διευκρινίσουμε καλύτερα, να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε τομείς που ανέφερε και ο Τζον. Σίγουρα μπορούμε να φωτίσουμε με το έργο μας περισσότερο τα πράγματα και αυτό αναφέρεται και σε σένα Σβέν. Με ξέρεις δεν κάνω πίσω στις δυσκολίες. Αν ε, δεν ε, έχουμε βάλει κάποια ουσιαστικά θέματα είναι γιατί ακόμα δεν τα έχουμε κλείσει. Όχι, αν δεν το έχεις πει αυτό που είπες δεν θα παρενέβαινα. Ε, είδαμε τα στοιχεία που δώσατε. Ε, τα δικά μας είναι λίγο διαφορετικά, αλλά δεν είναι προβληματικό αυτό. Είπα Προσπαθούμε να βρούμε λύση με το τέταρτο σενάριο. Είναι μια δυνατότητα. Θέλουμε να τα δούμε όλα αυτά συνεκτικά για να αποφύγουμε συνολικά, για να μην έχουμε παραπλανητικές πληροφορίες που σίγουρα δεν το θέλουμε. Αυτό ήθελα να πω. Η πρόθεσή μας είναι να εργαστούμε επικοδομητικά και να βρούμε λύση το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε την αξιολόγηση αυτής της ανταλλαγής των απόψεων. Ε, κατάλαβα ότι υπάρχει βούληση ε, συγκεκριμένη συνεργασίας ε, για εξέβρεση λύσεων που πρέπει να είναι λειτουργικές, αξιόπιστες, νομικά στέρες. Αυτή είναι η μόνη επιλογή για μας. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Καταλαβαίνω και ευχαριστώ τις ε, ε, διευκρινήσεις του κυρίου Μπερναντίνου και την Κομισιόν που είπε ότι δεν είναι η δεύτερη βέλτιστη. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει εφαρμογή της νομοθεσίας, συγκρισιμότητα, λεπτομέρειες που πρέπει να στηρίζονται σε νομοθεσία τέτοια ώστε να είναι αξιόπιστες για να έχουμε αξιόπιστη ενημέρωση των καταναλωτών. Πάνω σε αυτή τη βάση θα εργαστούμε και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορία επίσης που μάλλον θα λάβει χώρα μετά. Λοιπόν, τελειώσαμε το πρώτο κομμάτι, δηλαδή το σημείο 10 και πάμε στο 11 και πάμε στην ανταλλαγή απόψεων. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια και παρακαλώ τα μέλη ε, συνεχίζοντας τη συζήτηση να εστιάσουν όμως στο ψήφισμα και πώς αυτό θα συνταχθεί με τρόπο τέτοιο ώστε να ληφθούν υπόψη αυτά που είπαμε ο διάλογος, ε, η ανταλλαγή απόψεων σε αυτό το θέμα, ε, η βάση εργασίας και η ανάγκη να βρεθούν σαφείς απαντήσεις και βιώσιμες λύσεις στις ανησυχίες που εντοπίσαμε. Και η Κομισιόν και η ΕΙΟΠΑ ε, εργάζονται πάνω σε αυτό, αλλά δεν μπορούν να μας δώσουν ήδη από τώρα λεπτομέρειες σχετικά με την επίλυση αυτών των θεμάτων. Περβάνους. Αν θέλετε, μπορούμε να διακόψουμε και για πέντε λεπτά, δεν ξέρω, ή είστε έτοιμοι και μπορούμε να συνεχίσουμε αμέσως. αμέσως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΟΠΑ. Είναι συμπληρωματικές οι θέσεις τους και δεν ταυτίζονται. Είδαμε ταυτόχρονα ότι υπάρχει η πρόθεση να γίνει ό,τι χρειάζεται ούτως ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό σενάριο και έτσι να γίνει θέση σε ισχύ, να πραγματοποιηθεί με το αποφασιστέν χρονοδιάγραμμα. Θα πρέπει να συνεχιστεί η πίεση, ούτω ώστε να βελτιωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις, ούτως ώστε πρώτη πρώτου του 17 να τεθεί σε ισχύ αυτή η νομοθεσία. Αυτά. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι όπως έχουν τα πράγματα εμείς δεν δεχόμαστε αυτές τις κατεξοδότηση πράξεις και παραμένουμε πιστοί στο πνεύμα και το γράμμα των όσων αποφασίσαμε για το πρώτο επίπεδο. Οπότε και οι τροπολογίες 4 και 5 και ιδίως οι 5 θα πρέπει να αποτελέσουν vote και να τα βρουν από αυτόν οι πολιτικές ομάδες. Μετά έχουμε κάποιες παραγράφους στο αρχικό κείμενο του ψηφίσματος. Νομίζω ότι αυτές συγκεντρώνουν τη Γενική Συνένεση και οπότε με αυτή τη βάση θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την ε, συζήτηση μεταξύ της ε, ψήφισης για την ένστασή μας και της ψήφισης του κειμένου στην ε, Ολομέλεια. Αλλά υπάρχουν δύο συμπληρωματικά σημεία. Το πρώτο είναι το ότι θα πρέπει να θεωρούμε χρήσιμο να μνημονεύσουμε όπως και στην επιστολή που διαβιβάσατε πρόεδρε στον ε, Χίλ και στον Ντομπρόφσκης να υπάρχει λεγομνία για το Comprehensive Alert. Πρέπει, πρέπει να το πούμε. Και από αυτού υπάρχουν ε, δύο τροπολογίες. Οπότε τουλάχιστον για τη μία από αυτές τις δύο τροπολογίες να συμφωνήσουμε και να την εγκρίνουμε. Επίσης υπάρχει και το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Και σας ε, παραπέμπω στις τροπολογίες 15 και 16. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς ανώμα Σήμερα Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν θα τα καταφέρουμε και θα πρέπει να γίνει η αναβολή, γιατί όλοι λένε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το νομοθέτημα, τα νομοθετήματα και ότι θέλουμε το κείμενό μα να ολοκληρώσουμε την ε, εσωτερική αγορά, να υπάρξει των τον προϊόντων, να προστατεύσουμε τον ε, καταναλωτή. Οπότε για να κάτσουμε το βάλουμε κάτω, να ε, κάνουμε ό,τι χρειάζεται και όταν έρθει η ώρα τη ολομέλεια, σας ξανακάνουμε μια τροπολογία και να πούμε τότε, τότε, να πούμε ότι θέλουμε την αναβολή. Αλλά δεν είναι δυνατόν σήμερα να λέμε ότι θα πρέπει 100% να γίνει η αναβολή. Γι' αυτό σας λέω. Θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την πιο μεγάλη δυνατή πλειοψηφία. Μήπως μπορεί να απόσχει το ΕΛΚ ή να αποσύρει τις τροπολογίες 15 και 16. Ε, τότε θα έχουμε σίγουρα μια πολύ καλή αφετηρία για τις συνομιλίες και διαπραγματεύσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μην έχουμε τα ίδια το ίδιο πνεύμα όπως και σήμερα. Για τις τροπολογίες 15 και 16 θέλω να πω κάτι. Έχοντας ακούσει την Κομισιόν σήμερα και το θέμα second best επιλογή, πολιτικά μπορούμε να καταλήξουμε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί. Γιατί η πίεση θα πρέπει να διατηρηθεί έντονη. Χθες το βράδυ στα ΟΕΛΚ μιλήσαμε πολύ για αυτή τη στρατηγική διαδικασία και τι πρέπει να γίνει. Στην αρχή δεν ήμουν κι εγώ απόλυτα σίγουρος και ήμουν διατεθειμένος να ακολουθήσω τη λύση που προτείνει η Περβάνς. Αλλά διευκρινίζω, μετά από αυτά που είπε και ο Τζον Μπέργκεν για το second best, ότι ήδη γνώριζε ότι η Κομισιόν θα ακολουθούσε αυτό το δρόμο. Η διατήρηση λοιπόν των τροπολογιών είναι επιβεβλημένη και στο τέλος η διαπραγματευτική μας θέση ως κοινοβούλιο θα ενισχυθεί. Επαναλαμβάνω ε, αυτά που είπα στις δύο άλλες μου παρεμβάσεις. Ότι δηλαδή και εμείς σε τελευταία ανάλυση δεν θέλουμε αναβολή. Έτσι δεν είναι. Δεν θέλω όμως να καταλήξαμε σε χαοτική κατάσταση και η λεγόμενη λύση second best, δεύτερη καλύτερη, αυτό ε, κάνει, δυσχεραίνει τα πράγματα και στο τέλος θα καταλήξουμε σε ένα χάος. Κακό για όλους. Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Και σε τελευταία ανάλυση θα ψηφίσει η Επιτροπή. Αν άλλοι το βλέπουν διαφορετικά θα το δηλώσουν. Εμείς πάντως το δηλώνω ότι το ΕΛΚ δεν θέλουμε να, θέλουμε να αποφύγουμε το χάος μετά. Και τα λόγια της Κομισιόν με επιβεβαίωσαν, πρέπει να πω, στη θέση μου αυτή. Ευχαριστώ. Mr. Kamal. Thank you very much. Το ECR έχει συνυπογράψει δύο τροπολογίε. Η πρώτη κάνει αναφορά στην επιστολή που στείλαμε στην Κομισιόν, που ήταν αποτέλεσμα εσωτερικών διαπραγματεύσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είχαμε συμφωνήσει επί αυτής της επιστολής. Δεύτερον, ως σημείο κλειδί για το τι θέλουμε να αντιμετωπίσει η Κομισιόν ε, και χαίρομαι που συμφωνούν να διαπραγματευτούν μαζί μα. Το Δεύτερον, έχει σχέση με, την, με το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει μια διαφωνία για το χρονοδιάγραμμα και αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές θέσεις ε, για την ταχύτητα με την οποία μπορεί να προσαρμοστεί ο κλάδος κλπ. Ε, πάντοτε θα υπάρχουν κάποιοι που θα διαφωνούν με οποιαδήποτε νομοθεσία. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να τηρήσουμε τα όσα αναφέρει το νομοθετικό κείμενο επίπεδο 1 είτε συμφωνούσαμε είτε διαφωνούσαμε. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση αναβολή δεν σημαίνει ακύρωση της νομοθεσίας. Η αναβολή αφορά μόνο τις ε, θεμητές ε, επιφυλάξεις κάποιων που χρειάζονται περισσότερο χρόνο έτσι ώστε οι πληροφορίες που δίνουν στο κοινό να είναι σαφείς και ξεκάθαρες. Νομίζω ότι αυτό τέσσερις θα πρέπει να τις ακούσουμε πολύ προσεκτικά. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Jezek. Jezek. Ευχαριστώ. Το μόνο σαφές σήμερα είναι ότι ο κατεξουδότης κανονισμός της Κομισιόν θα πρέπει να απορριφθεί σήμερα. Ε, ορίζω την προθυμία της ε, Κομισιόν να ε, έργαστή, γοργά για να βρεθεί μια άλλη λύση. Όμως σήμερα δεν ακούσαμε καμία απάντηση από την Κομισιόν στις ερωτήσεις ουσίας. Οπότε είναι αδύνατον δύσκολο αυτή τη στιγμή να αξιολογήσουμε το επίπεδο στο οποίο θα εμφανιστούν δυσκολίες και διαφωνίες στο μέλλον. Η τροπολογία 16 ε, την οποία, ε, η οποία υποβλήθηκε και έχει παρόμοιο περιεχόμενο τη 14 την οποία είχαμε υποβάλει εμείς ε, ω εκτιμώντα. Επαναλαμβάνουμε δηλαδή εκεί ότι η διαπραγματευτική ομάδα θα πρέπει να ρωτήσει την Κομισιόν το, αν πιστεύει ότι θα πρέπει να αναβληθεί η θέση σε λειτουργία. Είτε έτσι είτε αλλιώ, όταν απορριφθεί ο κατεξοδότηση κανονισμό θα πρέπει να συνεργαστούμε, να συνέλθουμε, ε, να συνεδριάσουμε την Κομισιόν και να ε, δούμε ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα για την μελλοντική συνεργασία μας. Μακάρθη. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε προς τα που κινούμαστε. Εγώ προσωπικά θα ήθελα όλα αυτά να εφαρμοστούν το συντομό δυνατό, αλλά θα πρέπει να γίνει σωστά η εφαρμογή. η πράσινη ε, έθεσαν πολύ ε, ξεκάθαρα το πρόβλημα ε, με μια συγκεκριμένη ή ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή δεν δίδει το, αποτέλεσμα, το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα πρέπει το θέμα να αντιμετωπιστεί με τρόπο που θα ικανοποιήσει όλους έτσι ώστε να μην οδηγηθούμε σε περαιτέρω σύγχυση ούτε από πλευρά καταναλωτών, ούτε από πλευρά του κλάδου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συγγνώμη που είπα ΜΑΚ στο όνομα, μπροστά στο όνομά σας. Γίγολτ. Πρόκειται για συζήτηση που μοιάζει με συνάντηση συντονιστών ή σκιωδών ε, ε, ε, το θέμα ή, και με δημόσια διαβούλευση. Ε, ε, νομίζω ότι επί έχουμε δίκιο. Αν δεν συμφωνήσουμε σε ορισμένα σημεία κλειδιά, δεν χρειάζεται στην αντίρρηση που θα εκφέρουμε να πούμε ότι ε, χρειάζεται αναβολή. Ε, είμαι σίγουρος ότι η λύση θα μας δυσκολέψει. Οπότε ενδεχομένως θα χρειαστεί αναβολή. Παρ' όλα αυτά δεν χρειάζεται να το πούμε. Ε, αν είμαστε εδώ σκιώδεις ηγητές θα βρίσκαμε μια λύση και θα ήταν καλύτερο αυτό επί της ουσίας να ζητήσω από τους συναδέλφους να δουν τις τροπολογίες που έχουν υποβάλει επικοδομητικά ε, δεν είναι μεροληπτικές, ε, πιστεύω ότι αξίζουν τις υποστήριξη όλων. Τώρα υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στα δύο, στις δύο μεγάλες ομάδες για ένα σημαντικό σημείο και καλύτερα θα ήταν να το λύσουν μεταξύ τους πριν αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Ναι, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να λυθεί αυτό το θέμα. Το EFTD και το ENF και Φέρμπερ έχει το λόγο. Äh, Ευχαριστώ. Επειδή έκανα ε, μία από τις δύο προτάσεις ε, να ξέρουμε ότι ο κανονισμός PRIPS δεν λειτουργεί χωρίς την, νομοθετική, την κατεξουσιοδότηση πράξη. Οι εποπτικές αρχές πρέπει να ξέρουν τι κριτήρια πρέπει να ελέγχουν. Αλλιώς θα δημιουργηθεί μεγάλο αλαλούμ γιατί θα υπάρχουν διαφορετικές αρχές 27 διαφορετικοί επενδυτές σε 27 χώρες που θα λένε θα πρέπει να είναι περίπου έτσι, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν θα είναι γνωστό αφού δεν θα υπάρχει η κατεξουδότηση πράξη. Αν απορριφθεί, που άκουσα ότι είναι πιθανό, θα πρέπει να δούμε και τι συνέπειες θα επιφέρει η απόρριψή της. Χαίρομαι που βέβαια, ε, παρέμεινε ο κύριος Μπερναρντίνο, υπάρχει και η δυνατότητα μετά ο κύριος Μπερναρντίνο, που είναι ε, ε, ο επικεφαλής των τριών ρυθμιστικών αρχών, να πει ότι αφού ο νομοθέτης δεν μπορεί να λύσει το επίπεδο 2, θα το κάνω εγώ μέσα από ερωταπαντήσεις ή γνωμοδοτήσεις και τότε πάλι θα πρέπει να, εμείς να σκεφτούμε, μα συμφέρει κάτι τέτοιο. Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουμε τα πράγματα πρέπει να εξελιχθούν σύγχρονα και παράλληλα, αλλιώς δεν γίνεται. Παράκληση λοιπόν, αν μπορώ να επηρεάσω κατά την ομάδα S&D προς το συμφέρον όλων και των δυνητικών επενδυτών, των ιδιωτών επενδυτών, αυτών που ε, θέλουν να βάλουν στην αγορά τέτοιου είδους ε, δέσμες και προς το συμφέρον της εσωτερικής αγοράς που πρέπει να πάρει στο τέλος ένα ε, σωστά δομημένο πακέτο και όχι ένα πακέτο που θα ερμηνεύεται με 27 διαφορετικούς τρόπους. Γι' αυτό είναι σημαντικό το, level, ε, το επίπεδο 1 και το 2. Το level 1, το επίπεδο 1 δεν πρέπει να αλλάξει. Το έχουμε διαπραγματευτεί, συμφώνησα και εγώ. Αυτό ισχύει, δεν αλλάζει αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε να τεθεί σε ισχύ το επίπεδο 1 χωρίς το επίπεδο 2 και χωρίς να έχουμε χρόνο ούτως ώστε ο κλάδος να μπορεί να εφαρμόζει το επίπεδο 2 γιατί πρέπει και να εφαρμόζεται. Γι' αυτό παράκληση, τίποτα άλλο δεν λέει η τροπολογία μου 15, ε, τίποτα άλλο δεν λέει παρά να υποστηρίξετε αντίστοιχα το, το κείμενο. Ευχαριστώ. Would like Ευχαριστώ, Θες κάτι να προσθέσεις. Δεν είσαι υποχρεωμένη. Ωραία. Για να προχωρήσουμε. Να δούμε την ουσία. Είπαμε ότι τώρα πρέπει να ψηφιστεί το θέμα των αντιρρησιών μας και είπαμε ότι η ΟΠΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κινητοποιηθούν τόσο ώστε να καλύψουν το Κοινοβούλιο για αυτές του τις ε, ανησυχίες που πρώτον πρώτον επιμένει στο ότι στο πρώτο ε, επίπεδο θα πρέπει να τηρηθούν το γράμμα και το πνεύμα των συμφασίσαμε και επίσης αυτό το οποίο αναφέρθηκε στην ε, επιστολή που εσεί υπογράψατε πρόεδρε θα πρέπει αυτό να το εξετάσουμε με τα σοβαρότητα, διότι αντιλαμβανόμαστε τι λέει ο κύριος Μπερναρδίνο, ο οποίος ακόμα λέει ότι δεν έχει ολοκληρώσει όλα τα στοιχεία που θα πρέπει να απάντηση του και οπότε έτσι θα μπορούμε μεταξύ της σήμερα και της Ολομελίας να φτάσουμε σε κάποια λύση. Αλλά δεν θα πρέπει να λέμε θα το μελετήσουμε και θα δούμε και θα το κάνουμε. Γιατί αν μέχρι την ψήφιση δεν έχουν απαντηθεί όλα αυτά τα ερωτήματα, τότε δεν θα είναι δυνατόν να μπορέσουμε να ε, υποστηρίξουμε το RTS. Επίση, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το Comprehension Alert που για άλλη μια φορά ε, δεν καλύπτεται από το κείμενο. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε ούτω ώστε να εγκρίνουμε την σχετική τροπολογία, ούτω ώστε να μπει το κομμουνιστικό σε στο κείμενο. Ο καθένας επιμένει να αναλάβει τι ευθύνε του ε, για την λίστα ψηφορία. Αλλά σα ε, αναφέρω τα εξή τρία. Πρώτα πρώτα όσον αφορά τι τροπολογίε 15 και 16. Για αυτέ, ε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το ΕΛΚ εμένει στη θέση του. Και ο κύριο Φέρμπερ, ο μα είπε, μα εξήγησε γιατί εμένουν στο 15. Επίση, το 15, αποκλείει το 16. Άρα μια κομψήληση για όλους μας, ε, μέσα σε ένα πνεύμα συνεργασίας, ακριβώς όπως το επιθυμεί και η συνθήκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε ο κύριος Φέρμπερ να αποσύρει το 15. Και σε ανταλλάγμα είχαμε μια φορική τροπολογία επί του 16, το οποίο 16 θα συμπληρώνονταν ως εξής στα αγγλικά το 2016 θα γινόταν στο εξή. Απευθύνεται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτή την πρόταση για να αναβάλει την ημερομηνία θέσεω σε εφαρμογή του τάδε κανονισμού, τόσο ώστε να υπάρξει μια ομαλή εφαρμογή των όσων επιτάσσει ο κανονισμός και όσων επιτάσσει ο κατεξοδότη κανονισμός και, προφορική τροπολογία, να αποφευθεί η θέση σε ισχύ της νομοθεσίας πρώτου επίπεδου χωρίς το RTS. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένας εύστοχος αξιόλογος συμβιβασμός που θα συνοψίζει τα όσα συζητήσαμε σήμερα. Έχω και άλλα δύο προβλήματα όπως σας είπα και ελπίζω ότι θα υπάρξει ευρεία συνένεση στο Κοινοβούλιο. Πρώτα πρώτα να εγκρίνουμε την τροπολογία υπαριθμών 5, δηλαδή να υπενθυμίσουμε ότι εμείς δεν αμφισβητούμε την ε, νομοθεσία για το πρώτο επίπεδο που υπερψηφίστηκε από 600 και περισσότερο βουλευτές και κατόπιν να πάμε στο 11 και στο 13 για να καλύψουμε εκεί αυτό που θέλουμε για το Communication Alert να συγκεντρώσουμε ευρεία πλειοψηφία σε αυτές τις ε, ψηφίσεις και έτσι να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τις θέσεις δικές μας με την ΕΙΟΠΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος, είναι σαφές και θα διακόψουν τρογιά πέντε λεπτά για να πάμε μετά στην ψηφορία.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

Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στην ψηφοφορία. Καταρχήν δοκιμή. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πρέπει να ψηφίσουν πολλοί ακόμα. Ψηφίστε όλοι. Έχουμε 58, 57 ψήφισαν. Άλλος κλείνει η δοκιμαστική ψηφοφορία. Λοιπόν, το σχέδιο πρότασης ψηφίσματος για τα PRIPS. Α, τώρα έχουμε έναν S&D παραπάνω. Παράγραφος 1, αρχικό κείμενο, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Παράγραφος 2, αρχικό κείμενο, υπέρ, κατά, αποχές, παράγραφος 3, αρχικό κείμενο, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Τροπολογία 16 έχει αποσυρθεί. Έχουμε την προφορική τροπολογία και να ε, αποφύγουμε την εφαρμογή του επίπεδου 1 χωρίς τα RTS υπέρ. Κατά αποχές δεκτό, παράγραφος 4 αρχικό κείμενο υπέρ, κατά αποχές δεκτό, ε, αναφορικές ε, σκέψεις 1-2 υπέρ, κατά αποχές δεκτές, τροπολογία 1 υπέρ, κατά. Έλεγχος. Ελέγχουμε την τροπολογία ένα άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Αρχικό κείμενο, αναφορική πρόταση υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Αναφορική πρόταση 5 υπέρ ε, κατά αποχές δεκτό, τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 7 με 8 υπέρ κατά αποχές δεκτές, τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή, τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Απερίφθη. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Α, όχι. Έλεγχος. Γιατί σκεφτόμουν κάτι άλλο, τα, μετά. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 6 σε δύο μέρη θα, αν ένα από τα δύο γίνει δεκτά, αντικαθιστά όλο το κείμενο. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ναι, δεκτό. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Μαζί με τη 12. 9 και 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Το C, ε, αρχικό κείμενο, υπέρ κατά δεκτό, η αιτιολογική σκέψη C, δεκτή. D, αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Όχι, όχι, όχι, σαφώς, σαφώς, σαφώς, σαφώς εγκρίνεται, όχι. Ε, δεκτή. Αιτιολογική σκέψη C σε τρία μέρη, πρώτο μέρος, όχι δύο, δύο μέρη. Όχι, όχι, τροπολογία 10. Όχι, τρία είναι τα τμήματα. Πρώτο τμήμα της τροπολογίας 10, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος. Έλεγχος του πρώτου της 10. Πέρας. Απερίφθη. Τα υπόλοιπα καταπίπτουν. Ωραία. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 11. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος, αν και νομίζω ότι κατεψηφίστη. Άρχεται η ψηφοφορία. 13. Πέρας. Όχι, δεκτή. Η 14 είναι συμβατή υπέρ. Κατά αποχές Δεκτή. Τώρα ψηφ... Ορίστε κύριε Μπάλτς. Θα ήθελα ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Χρειαζόμαστε 16 μέλη για να γίνει αυτό, αλλά το ΕΛΚ είναι από πίσω από την πρόταση αυτή. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Βεβαίως. Τελικό κείμενο όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 55 υπέρ, κανείς κατά τρεις αποχές. Μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της απόρριψης αυτής της κατεξουσιοδότηση πράξης, λαμβάνοντας υπόψη και ε, ότι δεν, είναι, δεν υπάρχει πρίψ χωρίς αρτιές. Σαφές μήνυμα από το Κοινοβούλιο και τώρα θα αρχίσει γρήγορα ο διάλογος με την Κομισιόν. Η συγγήτρια όμως σίγουρα θέλει να πει κάτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλό την διαπραγματευτική ομάδα ε, υπό την ηγεσία των ε, συντονιστών ε, να συνέλθουν για να εντοπίσουν τα θέματα τα οποία θα χρειαστεί να διαπραγματευτούμε με την Κομισιόν. Μέχρι τώρα μιλούσαμε έτσι πολύ επίσημα και τυπικά επί της αρχής τώρα πολύ σύντομα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να εντοπίσουμε τα συγκεκριμένα σημεία ακριβώ στα οποία θεωρούμε ότι η Κομισιόν δεν εισάκουσε τις ε, ανησυχίες μας, έτσι ώστε να βρούμε λύση σε αυτά τα πολλά εκρεμή θέματα. Ευχαριστώ. Thank you very much. So, message is clear. We can move to the next vote. Σαφές. Περνάμε στην επόμενη, στο επόμενο θέμα. Προϋπολογισμός. Γνωμοδότηση. Συμβαστική πρόταση Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Έλεγχος, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Λίγη. Όχι. Ναι, λίγη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15. Υπέρ Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για τη 15. άρχιτε η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Υπέρ για τη 16. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επιβεβαίωση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές δεν βλέπω τους πράσινους ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η σοφορία λίγη σοφορία Απορρίπτεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική Β υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επιβεβαίωση. Λίγη φορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική D υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 45. Όχι, 46. Και 46. Θα πει 46 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Έχει καταπέσει μήπως αυτή. Ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο παρόλα αυτά. Παράγραφος 5 υπέρ. Κατά. Ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λήξη πληροφορία. Εγκρίνεται. 49. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά ηλεκτρονική σοφορία για την 57 άρχεται Λίγοι. Απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Λήξη ψηφοφορία απορρίπτεται. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 62. Υπέρ. Κατά. εποχέ. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. 43 υπέρ 7 κατά 6 εποχές. Συγχαρητήρια στον συγκητή. Περνάμε στις γραμμές του προπολισμού. Έκον 6, 4, 5, 7 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Έκον 64, 62 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Έκον 64-58 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 64-63 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 64-64 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 64-56 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 64-55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64-61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64-51 υπέρ κατά αποχές όχι, ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται Λίγη. Εγκρίνεται. Με μία ψηφοδιαφορά. Συμβαστική Α, πρώτη, ε, υπέρ. Κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική Β, υπέρ. απόχέ. αποχές, εγκρίνεται. 64-54, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64-53, με προφορική τροποποίηση, τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64-60 υπέρ κατά ηλεκτρονική επιβεβαίωση. Λίγη ψηφοφορία απορρίπτεται. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια στον εισηγητή ξανά. Κλείνουμε εδώ τη συνεδρίασή μας. Επόμενη συνεδρίαση Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 3 το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.